Συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και να εργαστούμε σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου δεν έχω. Οπότε πάμε κατευθείαν στο σημείο 2, αν δεν υπάρχει κανείς που να έχει κάτι να προσθέσει. ε, συγγνώμη, τρία. Έγκριση των πρακτικών. Είχαμε τη ε, πρακτικά από τις 24 ε, Σεπτεμβρίου, 13 Δεκεμβρίου και 10 Ιανουαρίου. Συμφωνείτε ότι μπορούμε να τα εγκρίνουμε αυτά πρακτικά. Δεν υπάρχει αντίδραση αρνητική. Άρα προχωρούμε στην έκθεση σε σχέση με τις συνεχιζόμενες διοργανικές διαπραγματεύσεις και εφόσον φτάνουμε το τέλος ε, της θετίας υπάρχουν πολλές ανεξελίξει ε, διοργανικές διαπραγματεύσεις που προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε Έχουμε λοιπόν το συντονισμό των ε, συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, ε, την εναρμόνιση της νομοθεσίας για την έκθεση για τα καρκινογόνα ε, τις καρκινογόνες ουσίες, πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές. Αυτό το ολοκληρώθηκε σήμερα και φτάσαμε σε αποτελέσματα. Έχουμε την οδηγία για τις διαφανείς και με συνθήκες εργασίας και δίνω το λόγο στους εισηγητές όσους είναι εδώ ώστε να μας κάνουν μια σύντομη ενημέρωση. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Κάζα για την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και ε, προσωπικής ζωής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως ίσως γνωρίζετε, το τελευταίο τριμερί για την ε, ισορροπία εργασίας ε, ε, ζωής ενημερώσαμε ότι τα κράτη-μέλη, ενημερωθήκαμε μάλλον, τα κράτη-μέλη θα δέχονταν την δίμηνη πατρική άδεια και ότι η ε, άδεια μητρότητας θα πληρώνεται στο ίδιο επίπεδο με την άδεια ασθένειας, την αναρωτική. Ενώ εμείς θέλαμε να καταβάλλονται περισσότερα ε, χρήματα. Σε σχέση τώρα με την το το μάκρος της σταδιοδρομίας ε, έχει σημασία, ενώ το Συμβούλιο έχει τη θέση να ε, υποβάλει την ε, τετράμινη γονική άδεια σε διάρκεια εργασίας ενός χρόνου και πάνω. Ενώ εμείς θέλαμε αυτό να ε, μπορεί να, γίνει, να ισχύσει νωρίτερα. Αυτό απορρίφθηκε από το Συμβούλιο. Το επόμενο τριμερή θα γίνει αύριο το απόγευμα και ελπίζουμε ότι θα είναι και ο τελευταίος. Έχω ένα καλό προέστημα. ότι αύριο θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση και για τα υπόλοιπα θέματα που δεν είναι τόσο κρίσιμα. Ευχηθείτε μου λοιπόν καλή τύχη για να έρθω με καλά νέα πίσω. Πραγματικά σας εύχομαι καλή τύχη και θα είμαι και εγώ παρούσα για να σας στηρίξω. Ε, Τώρα, ε, η συγγετής είναι ο κύριος Λέναρντ για την Λέναρντ. Ήρθατε στην κατάλληλη στιγμή, κύριε Λέναρτζ. Μπορείτε να μας ενημερώσετε σε ένα δίλεπτο, τρίλεπτο για την, αρχή, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ νόμιζα ότι θα μιλούσα μετά τον David Κάζα, οπότε λέω έχω χρόνο για να μπω μέσα, αλλά ήταν τόσο σύντομο, ήσουν τόσο σύντομο σήμερα David. Λοιπόν, ευχαριστώ. Ε, ψηφίσαμε στις 20 Νοεμβρίου για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας με καλή πλειοψηφία στην Επιτροπή Απασχόλησης αλλά και στην Ολομέλεια ε, αφού ε, αμφισβητήθηκε η εντολή και τα τρία θεσμικά όργανα είναι προσιλωμένα σε αυτή την υπόθεση. 8 ώρες ή λιγότερο μετά την ε, έγκριση της εντολής αρχίσαμε τον ε, τριμερή διάλογο επί Αυστριακής ακόμα Προεδρίας, αλλά και με παρουσία και της Ρουμανικής. Έχουν γίνει ήδη λοιπόν μερικές συνεδριάσεις στον τριμερή διάλογο, δεύτερη και τρίτη 8 ε, Ιανουαρίου και την περασμένη εβδομάδα στις 15 Ιανουαρίου πλέον επί Ρουμανικής Προεδρίας και η επόμενη συνεδρία είναι αύριο το βράδυ εδώ στις Βρυξέλλες. Βλέπετε λοιπόν ότι εργαζόμαστε με ταχύς ρυθμούς και με πολύ επικοδομητικό πνεύμα. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία για την ELA, ε, την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το πεδίο ε, που θα καλύπτει. Ελπίζω να καταλήξουμε ε, γρήγορα σε αυτό και σε ό,τι αφορά τους συνεννοημένους και κοινού ελέγχους, επιθεωρήσεις εργασίας μάλλον, και εκεί υπάρχει <clears throat> πρόοδος και προσπαθούμε να κατανοήσουμε ο καθένας τι θέλει από αυτή την υπόθεση και τι περιμένει. Υπάρχουν κάποια θέματα που εκκρεμούν ακόμα αλλά προχωρούμε, προχωρούμε. Για το ρόλο το διαμεσολαβητικό που θα έχει αυτή η αρχή και της ε, συμφιλίωσης και επίλυσης διαφορών, ποιος θα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο και ακόμα δεν έχουμε καταλήξει. Ε, αύριο θα αρχίσουμε να συζητούμε το ε, ρόλο του Γιούρες στην αρχή αυτή σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες που θα έχουμε στη λειτουργία στην αγορά εργασίας. 29 Ιανουαρίου και 5 Φεβρουαρίου έχουν προγραμματιστεί και νέες συνεδριάσεις ε, τριμερούς διαλόγου, άρα τηρούμε αυτό το πρόγραμμα που είναι πολύ σφιχτό και αυτό δεν θα μπορούσε να είχε καταστεί δυνατό χωρίς τη βοήθεια της Ορμανικής Προεδρίας ε, του Συμβουλίου και της δικής μας γραμματείας της Επιτροπής Απασχόλησης, την οποία πάντα ευγνωμονώ απείρως γίνεται καλή δουλειά, επικοδομητική και κανονικά θα πρέπει να προλάβουμε να τελειώσουμε πριν το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου την έκθεση αυτή που θα είναι και πολύ ευχάριστες ειδήσει, αλλά και θα αντανακλούν την ε, φιλοδοξία που είχαμε ως κοινοβούλιο θέση για αυτά τα θέματα. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο και προσβλέπω σε ταχεία ε, εκβασή και κλήρωση θετική φυσικά. Ε, προσπάθησα να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομος. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Ε, δεν βλέπω εδώ τον κύριο Μπαλάς και δεν ξέρω ποιος τον αναπληρεί, εάν τον αναπληρεί κάποιος. Α, έχουν αρχίσει οι τριμερείς διάλογοι και εδώ, θα επανέλθουμε. Τώρα, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και λοιπές ουσίες και έκθεσή τους στην εργασία. Έχουμε αυτή τη εβδομάδα ένα τριμερή διάλογο στον οποίο προεδρεύω εγώ για αυτό το θέμα. Η κυρία Ατζέα απουσιάζει επίσης, εξ όσων αντιλαμβάνω. Έχουμε και το σχέδιο κανονισμού για ένα κοινό πλαίσιο, οι ευρωπαϊκές στατιστικές. Σήμερα το χειριστήκαμε αυτό το θέμα και καταλήξαμε σε ένα καλό συμπέρασμα. Και θα το ολοκληρώσουμε, ίσως όχι τελείως τυπικά, αλλά ε, το μόνο που θα λείπουν θα είναι κάποιες υπογραφές. Και μετά έχουμε και την οδηγία για τις διαφανείς και προβλέψιμες συνθήκες εργασίας. Ε, και ο εισηγητής είναι ο κύριος Καλβέτ Σαμπόν, ο οποίος σήμερα στενεί και απουσιάζει και δεν μπορεί να μας ενημερώσει. Μπορώ όμως να σας πω ότι προχωρούμε και εκεί ε, πολύ καλά. Και η Προεδρία ίδια μας έχει βοηθήσει να προχωρήσουμε. Τούτων όλων λέχθεντων θα ήθελα να καλωσορίσω θερμότατα ε, τον Υπουργό και να του δώσω το λόγο. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης είναι ο κύριος Μπουντάη. Θα μας παρουσιάσετε την Ρουμανική Προεδρία μια εισαγωγή παρακαλώ, όχι πολύ μακροσκελή και μετά θα γίνουν ερωτήσεις και θα ακολουθήσει μια μικρή συζήτηση. Ελπίζω να συμφωνείτε. Θα πάρουν το λόγο οι συντονιστές των διαφόρων πολιτικών ομάδων σε ένα πρώτο γύρο και μετά οι υπόλοιποι, ε, υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Καλώς ορίσατε θερμά κύριε Υπουργέ και ε, πραγματικά προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας. Είναι τελευταίοι μήνες πριν τις εκλογές, αλλά πάρα πολύ έντονη και εντατική και ό,τι πετύχουμε μαζί θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και για ε, τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών στις ευρωεκλογέ, να τους κινητοποιήσει να ψηφίσουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικές εκλογές αυτές, ίσως οι σημαντικότερες ευρωεκλογέ όλων των εποχών από τότε που άρχισε η καθολική ψηφοφορία. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας και για τις εισαγωγικέ σας παρατηρήσεις. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 12 χρόνια μετά την προσχώρηση της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι από 1η Ιανουαρίου του 2019 εμείς έχουμε αναλάβει την ευθύνη να προεδρεύουμε στις εργασίες των ομάδων του Συμβουλίου της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για εμάς η Ρουμανική Προεδρία λοιπόν αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Είναι μια ευκαιρία εξαιρετική να αναδείξουμε τη σημασία που αποδίδουμε στις ευρωπαϊκές αξίες να επιβεβαιώσουμε και να υπογραμμίσουμε την ε, προσήλωσή μας στο ευρωπαϊκό ιδεώδες και να εργαστούμε για την περαιτέρω ενίσχυση του ευρωπαϊκού έργου. Αυτά είναι και το κέντρο βαρύτητας της Ρουμανικής Προεδρίας. Είναι τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω τους γενικούς στόχους της Ρουμανικής Προεδρίας αλλά και τις πιο συγκεκριμένες προτεραιότητες της επιμέρους που έχουμε ε, σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικών ε, υποθέσεων. Και ελπίζουμε όλα αυτά να τα προχωρήσουμε σε ικανοποιητικό βαθμό κατά το πρώτο εξάμεινο του 19 κατευθυντήρια γραμμή της Προεδρίας μας θα είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες, η έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας, του Ευρωπαίου πολίτη δηλαδή, με τις ανησυχίες και τις ανάγκες του. Θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι, αλλά, ε, αισιόδοξοι αλλά και ρεαλιστές. Αναγνωρίζουμε ότι με το Brexit εν εξελίξει και με τις ευρωπαϊκές εκλογές στον ορίζοντα, αλλά και με τη συζήτηση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τη συζήτηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, με όλα αυτά τα θέματα να τρέχουν, η Προεδρία μας δεν θα είναι μια κλασική Προεδρία και δεν θα αντιμετωπίσει μια κλασική ε, κατάσταση. Ωστόσο, είναι αταλάντευτη αυτή η προσήλωσή μας να βοηθήσουμε στο ευρωπαϊκό εγχείρημα και να συνεργαστούμε και σε επίπεδο Συμβουλίου αλλά και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε ρεαλιστές και να σημειώσουμε πραγματική πρόοδο στα θέματα που αποτελούν προτεραιότητά μας και έτσι να κομίσουμε στον Ευρωπαίο πολίτη απτά αποτελέσματα. Το μέλλον της Ευρώπης είναι ένα θέμα οριζόντιο που έχει να κάνει με όλες τις επιμέρους ε, πολιτικές. Και έτσι η σύνοδος του Σιβίου ελπίζουμε να αποτελέσει καθοριστικό σημείο, σημείο καμπή για την ενίσχυση του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Τέσσερις είναι οι πυλώνες γύρω από τους οποίους στρέφονται οι προτεραιότητές μας. Πρώτον, η Ευρώπη της σύγκλησης, δεύτερον, η Ευρώπη της ασφάλειας, τρίτον, η Ευρώπη ως ε, παράγων και δρόν οργανισμός σε παγκόσμιο επίπεδο και τέταρτον, η Ευρώπη των κοινών μας αξιών σε ό,τι έχει να κάνει με την Ευρώπη της σύγκλησης και με την Ευρώπη των κοινών αξιών, δηλαδή το πρώτο και το τέταρτο πυλώνα, η απασχόληση και οι κοινωνικές υποθέσεις καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος αυτών των πυλώνων και υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών θεωρούμε και επιθυμούμε να ισχύσει ο Ευρωπαϊκός Πυλώνας των κοινωνικών ή εργασιακών δικαιωμάτων, να έχουμε ίση πρόσβαση στην αγορά εργασίας, ίσες ευκαιρίες και βελτίωση των συνθηκών κοινωνικής συμπερίληψης, κοινωνικής ένταξης και καλύτερη κατανόηση και επικοινωνία μεταξύ ε, των ε, κοινωνικών παραγόντων όλα αυτά είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει σωστά και η εσωτερική αγορά, αλλά και για να λυθούν τα δημογραφικά προβλήματα διαφόρων χωρών μελών. Πρέπει να λύσουμε περισσότερα θέματα που έχουν να κάνουν με την κινητικότητα του εργασιακού δυναμικού, γιατί αυτό είναι παράγον αύξηση τη ανταγωνιστικότητα τη ευρωπαϊκή αγορά. Μα ενδιαφέρει ιδιαίτερω να καταπολεμήσουμε την αδήλωτη εργασία, αλλά και τι καταχρήσει που σημειώνονται σε αυτό το τομέα. Θέλουμε να υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα οργανισμό, μια υπηρεσία που να κομίζει προστιθέμενη αξία και που να δίνει και στους πολίτες και στις επιχειρήσεις και στη δημόσια διοίκηση το δικαίωμα για ελεύθερη πρόσβαση και ελεύθερη κυκλοφορία, έτσι όπως προκύπτει και προβλέπεται από τις συνθήκες, έτσι ώστε να μπορεί να κινηθεί καλύτερα και πιο ευέλικτα το εργασιακό δυναμικό. Θέλουμε να καταλάβουμε και να προστατεύσουμε τα κεκτημένα δικαιώματα των μεταναστών και των οικογενειών τους που αλλάζουν χώρα ε, για λόγους έβρεσης εργασίας και θέλουμε να προχωρήσουμε με το σχετικό κανονισμό ε, που προβλέπει τη σύσταση Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εργασίας. Θεωρούμε ότι η θέση των δύο συνομοθετών του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου είναι αρκετά ε, παραπλήσια. Στους τριμερείς διαλόγους προσπαθούμε να επιδιώξουμε τους ίδιους στόχους. Βλέπουμε ότι ε, ο στόχος είναι κοινό και για το Συμβούλιο και για το Κοινοβούλιο. Αποκλίνουσες απόψεις υπάρχουν στον τρόπο επίτευξης του ίδιου στόχου. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα κάνουμε το παν και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και ε, η πρόοδος ε, για τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των φύλων, ε, ευκαιρίες πρόσβασης και ανέλυξη στην αγορά εργασίας. Σε ό,τι έχει να κάνει με το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και προόνοιας, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Θέλουμε να προχωρήσουμε τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο και θέλουμε να αποδείξουμε ότι θα καταβάλουμε ως Ρουμανική Προεδρία κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση του φακέλου με τη λήξη της Προεδρίας μας να έχει ολοκληρωθεί. Θα προσπαθήσουμε σε κάθε περίπτωση το τελικό αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών. Γι' αυτό και στο Βουκουρέστι θα οργανώσουμε συνέδριο για το θέμα της κινητικότητας των εργαζομένων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ασφαλείς και ε, συνθήκες, ε, συνθήκες υγιεινής σε επαρκές ε, επίπεδο στο χώρο εργασίας. Η ασφάλεια και η υγεία στον χώρο εργασίας αποτελεί ένα πεδίο πολύ περίπλοκο. Οι πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ενδιαφέρονται και στοχεύουν προς αυτό το πεδίο και αποτελεί αυτό θεμελιώδες στοιχείο της αντίληψης που έχουμε για το πώς πρέπει να ρυθμίζεται μια αγορά εργασίας για να μην υπάρχουν, για να αποφύγουμε μάλλον ενδεχόμενες ε, στρεβλώσεις ε, και αποκλήσεις και για να μπορεί να γίνεται η δουλειά με αποτελεσματικό τρόπο. Άρα είναι σημαντικό να έχουμε συνθήκες εργασίας διαφανείς και προβλέψιμες. Και θα έχουμε όλα, όλα αυτά θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή δεν συμπίπτουν απολύτως οι θέσεις του Συμβουλίου με τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Το στόχος μας είναι όμως να φτάσουμε σε μια λύση που θα σέβεται τις πρακτικές που υφίστανται στα διάφορα κράτη-μέλη και συνάμα θα προάγουν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Σε ό,τι έχει να κάνει με την οδηγία για την έκθεση σε μεταλλαξιογόνε και καρκινογόνες ουσίες, σε αυτή την περίπτωση Σκοπός μας είναι να δείξουμε και να αναδείξουμε για άλλη μια φορά πόσο μεγάλη σημασία έχει για μας η ευημερία των πολιτών, η καλή διαβίωση των πολιτών. Οι συζητήσεις έχουν ε, διεξαχθεί, έχουν διεξαχθεί σε πολύ συνεργατικό πνεύμα μέχρι, στιγμή και θέλουμε, ε, μέχρι στιγμής και θέλουμε να εξάγουμε τα κατάλληλα συμπεράσματα πριν από τη λήξη της θητείας της Ρουμανικής Προεδρίας. Θα επαναλάβουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ασφάλεια και τις συνθήκες υγιεινής ε, στο χώρο εργασίας αλλά και στις νέες μορφές εργασίας και γι' αυτό θα οργανώσουμε συνέδριο και διάσκεψη για τους νέους πρακτικούς τρόπους με τους οποίους ε, γίνονται αυτές οι νέες μορφές εργασίας και πώς μπορεί να συσχετιστούν με την ασφάλεια και προστασία στο χώρο εργασίας η ισότητα των ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασία, η μείωση του μισθολογικού χάσματος, της μισθολογική απόκληση. η προαγωγή καλύτερη και βέλτιστης ισορροπία για την καλύτερη συμφιλίωση μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής είναι θέματα που μας ενδιαφέρουν η ισότητα ανδρών και γυναικών είναι απαραίτητο σπόρος για να φτάσουμε να κατακτήσουμε την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία η οποία θα συμπεριλαμβάνει όλους και η οποία ε, θα λειτουργεί αθρηστικά. Είναι πολύ σημαντικό να ενσωματωθούν τάχιστα οι σχετικές οδηγίες. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τη διαπραγμάτευση με το Κοινοβούλιο για την οδηγία που έχει να κάνει με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ε, προσωπικής οικογενειακής ζωής και θα επιδιώξουμε να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να ξεμπλοκαριστούν οι διαπραγματεύσεις, να βρεθεί ε, μια διέξοδος σε ό,τι έχει να κάνει με τη συζήτηση για ε, την ισορροπία ε, στις υψηλές θέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών, στις διευθυντικές ε, στελεχειακές θέσεις για τις επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Στις 15 Μαρτίου στο Αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών στις Βρυξέλλες και στα μέσα Ιουνίου στο Αρμόδιο Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τα θέματα αυτά και θα προσπαθήσουμε να υπάρξει συνεδρίαση Υπουργών Κοινωνικών Υποθέσεων στο Βουκουρέστι στις 10 και 11 Απριλίου του 19. Η ασφάλεια των εργαζομένων στο χώρο εργασίας είναι ένα θέμα που μας ενδιαφέρει και γι' αυτό θα οργανώσουμε και άλλα συνέδρια. Για παράδειγμα, ένα συνέδριο που να έχει να κάνει με τη συνεμετοχή των ανηλίκων και των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. 6 και 7 Μαΐου. Άλλο συνέδριο για τη βελτίωση και ε, αναβάθμιση των ε, δεξιοτήτων των ε, ε, ενηλίκων που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας 10 με 17 Μαΐου. Άλλο συνέδριο για την ισότητα ε, ε, ανδρών και γυναικών 29 και 30 Μαΐου. Μετά, νέος ορίζοντας και αλλαγή παραδείγματος στις 4, 5 και 6 Ιουνίου. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι και θεωρούμε ότι με την Προεδρία μας θα υπάρξουν αποτελέσματα απτά για τον Ευρωπαίο πολίτη. Εάν τα κράτη-μέλη μας βοηθήσουν, ε, και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας βοηθήσουν, πιστεύω ότι η Προεδρία μας θα είναι εξαιρετικά επιτυχημένη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση. Σας περιμένουμε με χαρά να σας υποδεχθούμε στη Ρουμανία φέτος το πρώτο εξάμεινο του 2019. Επομένως, σε ό,τι έχει να κάνει με το φάκελο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας, η Προεδρία καθορίζει τους στόχους της πρότασης αυτής. Να σας πω εν συντομία και μετά αν θέλετε με ρωτάτε. Εμείς θέλουμε να προχωρήσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις που είναι πολύ σημαντικές. Και το θετικό εδώ είναι ότι η θέση των δύο συνομοθετών είναι αρκετά παραπλήσια. Πολύ μικρά είναι τα σημεία, πολύ λίγα είναι τα σημεία στα οποία οι απόψει είναι αποκλίνουσε και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε τη σύγκληση κατά τη διάρκεια τη Προεδρία μα. Αυτά για αυτό το φάκελο. Τώρα για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλεια. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για το Συμβούλιο που πιστεύει ότι έτσι θα διευκολύνει την ελεύθερη κινητικότητα και κυκλοφορία των εργαζομένων μέσα από τον εξυγχρονισμό των συστημάτων κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια. Οι συνομοθέτε έχουν την ίδια φιλοδοξία, μοιράζονται την ίδια φιλοδοξία. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να προχωρήσει ο φάκελος αυτός ώστε το περισσότερο πριν από τη λήξη της θητείας της Ρουμανικής Προεδρίας. Τρίτον, η οδηγία για τη συμφιλίωση οικογενειακής και επαγγελματική ζωής στον τριμερή διάλογο αύριο. Είμαι σίγουρο ότι θα καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό, ένα εγχείρημα ιδιαίτερη σημασία, εξέχουσα σημασία για τον Ευρωπαίο εργαζόμενο και την οικογένειά του. Τέταρτον, συνθήκες προβλέψιμες και διαφανεί. Είχαμε ήδη τρεις τριμερείς διαλόγους κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας και θα προσπαθήσουμε, θα συνεχίσουμε αυτή την εντατική δουλειά για να εγκριθεί η οδηγία κατά τη διάρκεια της θητείας της Ρουμανικής Προεδρίας. Και τα δύο θεσμικά όργανα προτείνουν λύσεις ε, έτσι ώστε να υπάρξει σωστή ισορροπία. Και θεωρούμε ότι ο λόγος των, και ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων είναι κέριος κατά την εφαρμογή της οδηγίας. Θα πρέπει να διατηρηθεί αυτόν αυτονομία των κοινωνικών εταίρων, όπως ισχύει άλλωστε αυτό στα διάφορα κράτη-μέλη και ότι έχει να κάνει με το τέταρτο θέμα που μας απασχολεί, τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες στο χώρο εργασίας, Ξεκινούμε τους τριμερούς διαλόγους στις 16 Ιανουαρίου, τους ξεκινήσαμε όπως ξέρετε και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθούν διαπραγματεύσεις πριν από τη λήξη της θητείας της Ρουμανικής Προεδρίας για το Ταμείο προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και το σχετικό κανονισμό. Η πρόοδο που έχει σημειωθεί είναι αρκετή κατά τη διάρκεια τη Αυστριακής Προεδρίας κυρίω και η δικιά μας Προεδρία η Ρουμανική θα συνεχίσει προς την ίδια κατεύθυνση, θα πάρει τη σκητάλη από την Αυστριακή και ελπίζουμε ότι το Μάρτιο θα έχουμε καταλήξει σε μια ε, μερική γενική ε, συμφωνία ε, για το θέμα αυτό. Αυτά προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε ώστε να πετύχετε όσο γίνεται περισσότερο τους στόχους σας και εμείς τους δικούς μας. Έχουμε, ένα, Έχουμε ερωτήσεις, ε, παρεμβάσεις, πρώτα με τους συντονιστές και μετά με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Πρώτο ο κύριος Κάζα από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Υπουργέ για την ε, εισήγησή σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην ε, Προεδρία σας. Είναι μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή εφόσον πρόκειται για την τελευταία Προεδρία πριν το ηλίξη λήξη αυτής της θητείας. Έχουμε επιτάπητος σημαντικά θέματα που έχουν φτάσει σε κρίσιμη φάση. Γι' αυτό και χρειάζεται να έχουμε την υποστήριξη της Προεδρίας όσο γίνεται περισσότερο. διαφανείς και ε, σαφείς συνθήκες εργασίας, ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής, από ό,τι κατάλαβα είχα έτσι μια διέστηση ότι δεν είναι η μεγάλη σας αυτή η προτεραιότητα, αλλά εν πάση περιπτώσει εμεί έχουμε εργαστεί πολύ για αυτήν την οδηγία και είμαστε σε μια κρίσιμη φάση τώρα, βλέπετε. Και χρειάζεται να επιμείνουμε για να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Γιατί αυτή η οδηγία θα έχει μεγάλο αντίκτυπο στους πολίτες της Ένωσης. και μάλιστα ακόμη περισσότερο καθώς ε, η αγορά εργασίας κινείται προς πιο ευέλικτες μορφές εργασίας και γι' αυτό και θα πρέπει να προσέξουμε αυτά τα σημεία ειδικά για τις γυναίκες. Ελπίζουμε λοιπόν να διατηρήσετε την έμφαση ε, που θέλουμε για αυτό το θέμα. Τώρα, για τα δύο ταμεία. Και το κοινωνικό, το ταμείο και το ταμείο για την παγκοσμιοποίηση. Είμαστε κάπως απογοητευμένοι και για τα δύο αυτά και ελπίζω ότι θα μου πείτε κάποια πράγματα αργότερα. Ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η κατάσταση. Πώς θα βρείτε λύσεις. Γιατί το να μην έχετε κάποια θέση δεν είναι πολύ ευχάριστο. Σας ευχαριστώ κύριε Κάζα και τώρα δίνω το λόγο ε, στην συντονίστρια των Σοσιαλιστών, την κυρία Γιονγκέριους. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και σας ευχαριστώ Υπουργέ που ήρθατε ε, και μας κάνατε την εισήγησή σας για τις ε, προτεραιότητές σας. Μου αρέσει, θα πρέπει να πω, ο συνδυασμός μιας ρεαλιστικής και φιλόδοξης προσέγγισης, διότι νομίζω πως η φιλοδοξία είναι αυτό που χρειαζόμαστε εάν θέλουμε να ε, ολοκληρώσουμε κάποια από αυτά τα σημαντικά θέματα που είναι ε, τώρα ε, προς Σας ευχαριστώ λοιπόν που είστε ρεαλιστής αλλά και φιλόδοξος μαζί για την ολοκλήρωση αυτών των τριμερών. Πιστεύω και επίσης είμαι πολύ ευτυχής που τονίσατε την ανάγκη σύγκλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι επίγουσα η κοινωνική και οικονομική συνοχή στην Ένωση και πρέπει να σας πω ότι η συζήτηση για το Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο της ε, Συνοχής ε, είναι θέματα τα οποία επίσης χρειάζονται ε, αντιμετώπιση και γι' αυτό περιμένω την απάντηση που θα δώσετε στο συνάδελφο Κάζα. Είμαι Ε, ευτυχής για τις προτεραιότητες που αναφέρατε. Δεν θέλω να, να, περιπλακούν τα πράγματα στους συνεχιζόμενους τριμερείς, γιατί ξέρω πως πολλοί έχουν ασχοληθεί πολύ περισσότερο από ότι εγώ. Θα ήθελα όμως να χρησιμοποιήσω αυτή την ευκαιρία για να πω ότι δεν πιστεύω ότι η έδρα ε, θα είναι η πρώτη πρώτη προτεραιότητα. Θα ήταν καλύτερο να μπει σε μια τροχιά η υπόθεση αυτή και να ασχοληθούμε με το θέμα της έδρας αργότερα. Ε, ώστε να δούμε πού θα είναι, ποια θα είναι η έδρα της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Καταπολέμηση της, ε, των ε, παραβάσεων, των καταχρήσεων επίσης είναι πολύ σημαντική ε, γιατί αυτό είναι προς όφελος των εργαζομένων. Τώρα, εάν είστε αρκετά φιλόδοξοι, όπως και ο συνάδελφός μου, ότι θα ολοκληρωθεί αυτός ο τριμερής αύριο, τότε θα είναι πολύ θετικό αυτό για την ισορροπία μεταξύ εργασιακής και προσωπικής ζωής. Επίσης, διαφανής ε, και σαφείς ε, συνθήκες εργασίας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους εργαζόμενους άνδρες και γυναίκες της Ένωσης. Δείτε για παράδειγμα εκείνες τις, ε, τις γυναίκες που εργαζόνται στον τομέα της υγείας με τα ευέλικτα συμβόλαια εργασίας θα πρέπει να ισχύουν ε, ε, στέρεοι κανόνες για να μπορούν να έχουν ισορροπία στη ζωή τους αλλά και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για να δημιουργηθεί βεβαιότητα για τους εργαζόμενους στην υγεία. Ήλπιζα επίσης ότι θα σημειωθεί πρόεδρος για τα καρκινο, ε, τους καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες ουσίες γιατί ε, και αυτό θα σήμαινε πως οι εργαζόμενοι θα εργάζονται ε, με ασφαλή τρόπο και θα φτάσουν ε, στα γεράματα υγιής. Και τέλος, αν όντω έχετε ολοκληρώσει το κοινό πλαίσιο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές σήμερα το πρωί, ορίστε ένα θέμα που βγαίνει από τη φιλόδοξο κατάλογο και πραγματικά σας συγχαίρω που ολοκληρώσατε ήδη αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. του, συντονίστρια του ECR, κυρία Μάκινταερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και σας, Υπουργέ, που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας. Κληρονομήσατε την Προεδρία σε καιρούς πάρα πολύ έτσι, φορτωμένος. Η Πρωθυπουργό σα όμω, που είναι και πρώην Ευρωβουλευτή, ξέρει ε, τι γίνεται ε, και από τα μέσα πώ γίνονται οι διαπραγματεύσει και πώ μπορούν να συνεργάζονται οι συνομοθέτες. Ακούσαμε τι προτεραιότητε σα, τι νομοθετικέ, που καλύπτουν σχεδόν πάντο επιστητών. ακούσαμε και τους άλλους συντονιστές να βάζουν ε, όλα τα θέματα σε ύψιστη προτεραιότητα. Μα μπορεί να είναι όλα τα θέματα ύψιστη προτεραιότητα. Η δική μου προτεραιότητα είναι να είναι καλή νομοθεσία. Um, Η ομάδα μου ε, ήταν ο πρωταθλητής για την καλύτερη νομοθεσία, το F νομοθετή, είναι αυτό το Better Regulation, για τη Διοργανική Συμφωνία. Είναι για μας η πρώτη προτεραιότητα. Πόσο πιστεύετε ότι θα μπορέσουν οι συνομοθέτες να παράγουν καλή ποιοτική νομοθεσία για τους Ευρωπαίους πολίτες που να μπορεί να εφαρμόζεται και να έχει αποτελέσματα επί τόπου. Θα συμφωνούσατε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία να καταλήγουμε σε καλή νομοθεσία παρά να τα ολοκληρώσουμε όλα και να τα ξεπετάξουμε πριν τελειώσει η θητεία μας, οπωσδήποτε για να κλείσουν. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο των ε, φιλελευθέρων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας. Λέει η κυρία Τόμ. Δυστυχώς ε, ασθενεί ο κύριος Καλβέρης Σαμπόν, ο δικός μας συντονιστής και μιλώ εγώ στη θέση του. Και για μας είναι προτεραιότητα η ισορροπία του εργασιακού και του ιδιωτικού βίου, και δική σας προτεραιότητα. Έχετε και ελπίζουμε φιλόδοξη νομοθεσία που θα έρθει πριν το τέλος της θητείας για να προάγουμε την ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας. Και η δική μου ομάδα, φιλελεύθερη, καλούμε τη Ρουμανική Προεδρία να κάνει ό,τι μπορεί ε, για να προχωρήσουν αυτά τα θέματα και ε, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας μέχρι το τέλος κοινοβουλευτικής περίοδου. Η διευκόλυνση της κινητικότητας των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η άρση των εναπομεινάντων ε, φραγμών και εμποδίων είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας για να μπορούν οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθερα. Η αναθεωρημένη πρόταση για τον κανονισμό, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ε, αυτό ακριβώς έχει ως γνώμονα θα πρέπει να διευκολύνουμε τις διαδικασίες για τη φορητότητα ή τη μεταφορά των συνταξιωτικών ε, και άλλων δικαιωμάτων που έχουν θεμελιώσει οι πολίτες που εργάζονται σε άλλη χώρα. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να ε, επιταχύνουν στην ατζέντα και το θεματολόγιο για τις νέες δεξιότητες, για την καλύτερη κατάρτιση και νέες δεξιότητες μεταξύ αυτών και ψηφιακές δεξιότητες για την ενίσχυση της απασχόλησης. Έχουμε και το θέμα της διαβίου μάθησης, της μετεκπαίδευσης, του παρακαθορισμού των δεξιοτήτων και της απόκτησης δεξιοτήτων για να ε, αρθούν οι αναντιστοιχίες που βλέπουμε στην αγορά εργασίας. Επίση, οι φιλελεύθεροι λυπούνται που ε, είναι ακόμα εμπλοκή στο Συμβούλιο η διαδικασία των διακρίσεων και η σχετική οδηγία. Ελπίζουμε ε, η δική σας Προεδρία να το προεθήσει αυτό το θέμα. Τα κράτη-μέλη πρέπει να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για τη συμπερίληψη ατόμων με αναπηρίες στην αγορά εργασίας, ε, έροντας τους νομοθετικούς φραγμούς και τα εμπόδια και προσαρμόζοντας τους χώρους εργασίας για την φυσική πρόσβαση των ΑΜΕΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. GoNGL. Αποσιάζει Γκουε. Προχωρούμε στους πρασίνους. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τη Ρωμανική Προεδρία και βλέπω ότι οι προεδρίες από μικρότερες χώρες φέρνουν πολύ καλά αποτελέσματα. I think in your presentation... Ε, στην παρουσίασή σας είπατε ε, ότι είχατε δύο τμήματα. Ε, έγινε σε δύο μέρη χρονικά η Προεδρία. Πρώτο όλα αυτά τα νομοθετήματα που έχουμε και μετά η περίοδος προς τις εκλογές και μετά τις εκλογές. Ένα από τα θέματα που συνδέουν και τα δύο είναι η ελεύθερη κυκλοφορία. Ε, τώρα εμείς εργαζόμαστε για θέματα κοινωνικής ασφάλισης ε, και ε, Επειδή είμαι και από το Ηνωμένο Βασίλειο, συμπτωματικά, εγώ είδα πόσο σημαντική ήταν η ελεύθερη κυκλοφορία και πόσο ευεργετική ήταν για την οικονομία μας και τον τρόπο με τον οποίο υποφελήθηκαν οι δικοί μας πολίτες ε, ε, που διαβιούν εκτός ε, του Ηνωμένου Βασιλείου αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτά τα πράγματα είναι αμοιβαία. Καμιά φορά όμως προβάλλονται ως εντάσεις μεταξύ των Ανατολής Δύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας, εσείς έχετε την πρόθεση να βοηθήσετε για την αμοιβαία κατανόηση και να του πείσετε όλους ότι είναι προ όφελο όλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και δεν σημαίνει ότι κάποιες χώρες εκμεταλλεύονται ε, τις άλλε για, ε, για ίδιο όφελος α πούμε. Πώς μπορεί η Προεδρία σας να συνεισφέρει ε, σε αυτή την αμοιβαία κατανόηση. Και για να αναφερθώ σε κάτι άλλο για το θεματολόγιο σχετικά με τις δεξιότητες, ε, η δική μας Επιτροπή έχει ε, κάνει πάρα πολλή δουλειά για να δούμε πώς μπορεί η αγορά εργασίας να ανταποκριθεί στις κλιματικές αλλαγές, στην ενεργειακή αποδοτικότητα. Όλα αυτά ε, θα τα εντάξετε στη διάσκεψη που μας είπατε ότι θα γίνει για τις δεξιότητες. Η FTD απουσιάζει από ό,τι βλέπω. Οπότε η ομάδα ENF επίσης απούσα. Περάσουμε μέσα στο δεύτερο γύρο των υπόλοιπων μελών που ζητούν το λόγο. Ο κύριος Πάβελ πρώτος. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, bine ați venit în Parlamentul European. Mă bucur să vă văd. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ που είστε εδώ και που μας παρουσιάσατε τις προτεραιότητες για την πρώτη Ρουμανική Προεδρία. Εμείς νιώθουμε πραγματική υπερηφάνεια και θέλουμε να αποδείξουμε ότι μπορούμε να είμαστε φιλόδοξοι. Παρόλο που είμαστε και ρεαλιστική, γιατί η Ρουμανική Προεδρία δεν θα κρατήσει μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν πρέπει να είμαστε μόνο ρεαλιστές, όμως πρέπει να είμαστε και αισιοδόξοι και πολύ καλά το κάνετε. Ε, η Μαρία Ζωά η Συνάδελφό μου, δεν είναι εδώ παρούσα αυτή τη στιγμή. Όμω αυτό το θέμα του κοινωνικού πυλώνα, του Ευρωπαϊκού, ευρωπαϊκού κοινωνικού πυλώνα, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την πολιτική μου ομάδα. Πρέπει να παρουσιάσουμε αυτά αποτελέσματα στου πολίτε και η φιλοδοξία που επιδεικνύεται ε, μα κάνει να σκεφτόμαστε και να αισιοδοξούμε ότι πράγματι θα καταλήξουμε σε αυτά αποτελέσματα. Ο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό πυλώνα είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Εσεί έχετε ένα Υπουργείο που ε, ονομάζεται διαφορετικά από την ε, κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Εσείς έχετε Υπουργείο Κοινωνικής Δικαιοσύνης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Έτσι είναι ο τίτλος ε, στα, ε, στο Ρουμανικό Υπουργείο και ελπίζουμε η Ρουμανική Προεδρία να συμβάλλει στην κοινωνική δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή ε, Είναι η έβδομη χώρα από πλευρά πληθυσμού και όταν φύγει το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι η έκτη χώρα από πλευρά πληθυσμού. Δυστυχώ όμω για τη ρουμανική οικονομία, 4 εκατομμύρια Ρουμάνοι δεν ζουν στην ρουμανική επικράτεια, ζουν και εργάζονται σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω δεν είμαστε μικρή χώρα, είμαστε η 7 από πλευρά πληθυσμού και θα γίνουμε πολύ σύντομα και η έκτη. Ποια είναι τα μέτρα που σκοπεύετε να πάρετε έτσι ώστε να επιστρέψουν και οι Ρουμάνοι πολίτε στην Ρουμανία να εργαστούν στη χώρα του, γιατί μα λείπει εργασιακό δυναμικό. Και εσείς ε, και άλλοι υπουργοί έχουν μιλήσει για υποτροφίες εργασίας, γιατί χρειαζόμαστε ε, ε, εργασιακό δυναμικό. Ναι επιστρέψουν οι Ρουμάνοι που έχουν φύγει. Σε κάθε περίπτωση θα σε ευχόμαστε καλή επιτυχία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είπε ότι δεν θα, ε, δεν θα διαπραγματευτεί για περισσότερες από 5 ή 6 εβδομάδες και μέσα σε αυτές πρέπει να καταλήξετε σε όλες σας τις προτεραιότητες. Η κυρία Λόπε Φοντανιέ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίσατε κύριε Υπουργέ. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι πολύ σημαντικό για εσάς να έχετε επιτυχία, αλλά και για τον Ευρωπαίο πολίτη να στεφθεί το έργο σας με επιτυχία. Το σημαντικό είναι να καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι σημαντικό να καταλάβει ο Ευρωπαίος πολίτης ότι ο κοινωνικός πυλώνας είναι προτεραιότητα για εμάς, είναι προτεραιότητα για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην νιώθει ότι αυτά είναι θέματα παραμελημένα. Όπως είπε και ο συντονιστής, την ε, ε περασμένη εβδομάδα εγκρίναμε με ευρεία πλειοψηφία τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΣΥΝ, Θα χαρακτηρίσει την περίοδο 2021-2027 ενδιαφέρει άμεσα τον Ευρωπαίο πολίτη, έχει άμεσο και θετικό αντίκτυπο στο εκπαιδευτικό σύστημα, στο σύστημα κατάρτισης των κρατών μελών, άρα και στην αγορά εργασία την εθνική στη συνέχεια στι ε, διάφορες χώρες και έτσι βοηθάει στην ε, συμμετοχή, την ένταξη στην κοινωνία των πιο μειονεκτικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σε κάθε περίπτωση αυτό συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με τις προτεραιότητες της δικής σας Προεδρίας της Ρουμανικής. Μιλήσατε για τις δημογραφικές εξελίξεις και αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ισπανία, το πληθυσμιακό. Όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε συμπεριλαμβάνονται στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Άρα δεν είναι κατά το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή θεώρησε ότι πρέπει να ασχοληθούμε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλες οι πολιτικές ομάδες κατέληξαν σε συμφωνία για να εγκρίνουμε με ευρία πλειοψηφία το σχετικό κανονισμό. Και νομίζω ότι μιλώ εξ ονόματο όλων των πολιτικών ομάδων όταν λέγω ότι είναι ένα θέμα προτεραιότητα, είναι ένα θέμα που πρέπει να μα απασχολήσει και προσπαθήσαμε να δώσουμε ένα υπόδειγμα, ένα παράδειγμα στον Ευρωπαίο πολίτη ε, καλής ευρωπαϊκής πρακτικής. Επομένως, ποια είναι η άποψή σα για τη σημασία που δίνει η δική σα Ορμανική Προεδρία για την έκθεση αυτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που έχετε θέσει υπόψη σα και εμά είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό. Είναι σημαντικό, θα είναι ένα σωστό και καλό και θετικό μήνυμα που θα στείλουμε στον Ευρωπαίο πολίτη. Εμείς ως Κοινοβούλιο κάναμε το κομματάκι που μας αναλογεί, κάναμε τη δουλειά που μας αναλογεί, περιμένουμε και το Συμβούλιο να πράξει το ίδιο. Ε, Πρέπει να ξεχάσουμε τους μαξιμαλισμούς και τέτοιου είδους πληθωριστικές προσεγγίσεις, αντιθέτως να καταλήξουμε σε μια ισορροπημένη συμφωνία την οποία να μπορούν να στηρίξουν όλες οι πολιτικές ομάδες. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας εύχομαι κάθε επιτυχία για την ε, Ρουμανική Προεδρία. Έχετε βαρύ έργο. Η Προεδρία σας διαρκεί έξι μήνες, όπως όλες οι Προεδρίες, αλλά αντιμετωπίζει πολύ σημαντικές προκλήσεις. Πρώτη είναι να κλείσετε τις τελευταίες διαπραγματεύσεις και ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι διαπραγματεύσεις. Έχουμε δουλέψει πολύ για την κοινωνική Ευρώπη. Εσείς φέρετε τώρα την ευθύνη να ολοκληρώσετε τα κείμενα που έχουμε δουλέψει. Θα ήθελα να βάλετε όλο σας ε, το πάθος και την αποφασιστικότητα για να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις γιατί πρόκειται για πολύ ουσιαστικά κείμενα που θέλουμε οπωσδήποτε να ολοκληρωθούν. Αυτό είναι ο δικό σα καθήκον. Το δεύτερο σα καθήκον είναι ότι οι Ευρωπαίοι πολίτε πρέπει να αισθανθούν ότι η Ευρώπη δουλεύει για εκείνου. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να έρθει κοντά η Ευρώπη στον πολίτη, να τον καταλάβουν στη διάρκεια των εκλογών κυρίω και αυτό είναι στη διάρκεια τη Προεδρία σα που θα γίνει, πολύ βαριά ευθύνη, δεν είστε μόνοι, όλοι είμαστε γύρω σας, κοντά σας αλλά τυχαίνει η Ρουμανία μια νέα χώρα εισερχόμενη και που παίρνει για πρώτη φορά την Προεδρία έχει το καθήκον να δείξει πως η κινητοποίηση ή υπερευρωπαϊκή, φιλοευρωπαϊκή θα πρέπει να είναι το η εικόνα μας για το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι τεράστια ευθύνη γιατί είναι όλη αυτή η δουλειά της επόμενης θητείας. Όλες οι συνθήκες και όροι εργασίας της επόμενης θητείας εξαρτώνται από αυτό, από αυτή σας τη δέσμευση. Σας εμπιστεύομαι, αλλά μην το ξεχνάτε. Υπάρχουν επίσης κάποια σημεία που εμένα μου είναι πολύ ε, αγαπητά. Μιλήσατε για ισότητα ανδρών γυναικών και είπατε ότι θέλετε να καταργήσετε το χάσμα μεταξύ, αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αν εσείς τα καταφέρετε μέσα σε έξι μήνες, εγώ θα πάω να ζήσω και να εργαστώ στη Ρουμανία. Είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο. Αλλά θέλω να σας πω πάνω απ' όλα ότι πέρα από το χάσμα το μισθολογικό θα πρέπει να επιτεθείτε και στο θέμα της γυναικείας σταδιοδρομίας και θέλω να επιμείνω σε αυτό γιατί στις προεκβολές και η συνάδελφος Τζιν Λάμπερτ πολύ ωραία το είπε για τις νέες απαραίτητες ε, δεξιότητες αλλά γνωρίζουμε ότι στη βάση της πυραμίδας των ε, θέσεων απασχόλησης 15% των θέσεων θα καταργηθούν τα επόμενα χρόνια. ή ε, Θα είναι οι θέσεις χαμηλών προσόντων. Δυστυχώς είναι θέσεις εργασίας όπου οι γυναίκες είναι πιο πολυάριθμες από τους άντρες. Εάν λοιπόν δεν ασχοληθείτε τόσο με την αναγνώριση των δεξιοτήτων των γυναικών όσο και της δυνατότητας κινητικότητας στη σταδιοδρομία από το πιο χαμηλό σημείο μέχρι την κορυφή της πυραμίδα γιατί ο στόχος δεν είναι να έχουμε μόνο περισσότερες γυναίκες σε διευθυντικές θέσεις πρέπει να βάλετε όλες αυτές τις αρμοδιότητες και τις νέες αρμοδιότητες στην υπηρεσία κινητικότητας όλων των ε, υπαλλήλων στην Ευρώπη αλλά κυρίως για τις γυναίκες γιατί είναι εξαιρετικά ευαίσθητο το θέμα για τις γυναίκες και δεν είναι θέμα ισότητας ανδρών γυναικών αν και είναι και αυτό είναι ένα θέμα που αφορά την φτωχοποίηση των γυναικών και αυτό είναι πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό θέμα Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα ήθελα ανάμεσα στα εργοτάξια τα οποία εσείς θα ξεκινήσετε εδώ να ε, επιταχύνετε στο συγκεκριμένο θέμα. σε ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Σόγκορ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία κατά τη διάρκεια ε, του σύντομου διαστήματος. Ένα τρίμηνο είναι ουσιαστικά που θα έχετε την Προεδρία. Θέλω να κάνω μια ερώτηση ε, για τον κλάδο των μεταφορών που απασχολεί όμως εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους, ιδιαίτερα ε, στις παρυφές της Ευρώπης. Οι δέσμοι για την κινητικότητα που αφορά τις οδικές μεταφορές ε, έχει να κάνει και με την εσωτερική αγορά. Και όπως γνωρίζετε μετά από δύο απόπειρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν εγκρίθηκε η δέσμη αυτή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθαθέσει κάποιες προτάσεις που τις θεωρεί πακέτο, δέσμη. Εσείς στο Συμβούλιο συμφωνείτε με αυτή την προοπτική. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο μας, τον κύριο Κλοντ ε, Γολά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Πραγματικά ενδιαφέρον ε, είναι ο άξονας στον οποίο βασίζεται την Προεδρία σας, που είναι ο πολίτης. Ο πολίτης είναι το σημαντικότερο. Καθημερινά αυτό διαπιστώνουμε ότι υπάρχει απόσταση και θα πρέπει να συμφιλειωθούν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, οι ευρωπαϊκές διαδικασίες και και με τον Ευρωπαίο πολίτη. Πώς θα γίνει αυτό. Ο καλύτερος τρόπος είναι να το κάνουμε όσο γίνεται πιο συγκεκριμένα και να απαντάμε στα μελήματα των πολιτών, στα προβλήματά τους, στην καθημερινότητα. Τα κοινωνικά, τα θέματα απασχόλησης είναι συγκεκριμένα, είναι άμεσα, είναι ανθρώπινα θέματα. Ε, και σας συγχαίρω γι' αυτό. Σημειώνω ότι στην εισαγωγή σας ε, ε, ε, μιλήσατε σε παράλληλους πυλώνες. Από τη μια έχουμε τη φιλοδοξία, από την άλλη έχουμε το ρεαλισμό. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να σας απαντήσω ότι ο ρεαλισμός σήμερα σημαίνει να είσαι φιλόδοξος. Δηλαδή ακριβώς να είσαι ρεαλιστής σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, επιτρέψαμε να αφερθώ σύντομα σε δύο πράγματα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα ε, βαθιά δημοκρατικό. Έχουμε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, η οποία όμως για να λειτουργεί σωστά θα πρέπει να συμπληρώνεται από ε, όργανα ε, κοινωνικής διαμεσολάβησης. Οι εργοδοτικές οργανώσεις, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων είναι τέτοια σώματα που μεσολαβούν. Εσείς θα πάρετε τέτοιες πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση των κοινωνικών εταίρων για να μπορέσουν να συμμετέχουν στην εξέβρεση των συγκεκριμένων απαντήσεων που χρειαζόμαστε. Ένα δεύτερο στοιχείο που απασχολεί και την πρόεδρο και εμένα για τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες οσίες είναι πάρα πολύ σημαντικό γι' αυτό και πολύ συγκεκριμένο. Μα τι πιο συγκεκριμένο επιτέλους για τον κόσμο από την υγεία του. Τι υπάρχει πιο συγκεκριμένο να ξέρουν ότι αύριο δεν θα χάνουν τη ζωή τους, την θα καταστρέφουν την υγεία τους πηγαίνοντας στη δουλειά τους. Ακριβώς εδώ διασταυρώνεται αυτό με τη δική σας φιλοδοξία. Και ακούμε ένα σλόγγαν το τελευταίο καιρό, η Ευρώπη που προστατεύει. Εδώ λοιπόν η ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να προστατεύει τους πολίτες. δεν χρειάζεται ένα τρίτο πακέτο τώρα, ας πούμε, ή μια τρίτη φάση. Ε, μπορεί στην ε, δική σας Προεδρία να ολοκληρωθεί η δεύτερη ενότητα και βλέπουμε από εκεί και πέρα. Και τέλος, νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να γίνει στη δική σας Προεδρία, αλλά και στην επόμενη, γιατί είστε σε λίγο μεταβατική Προεδρία, για την αναθεώρηση αυτής της οδηγίας για τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες, δεν θα πρέπει να περιορίζεται ε, πρώτη φάση, δεύτερη φάση, τρίτη φάση και αύριο τέταρτη. Θα πρέπει να είναι μια διαδικασία πάγια και διαρκής, γιατί είναι εκατοντάδες, χιλιάδες ουσίες, εκατομμύρια με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι και εκτίθενται οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους αυτές. Και κάθε τρεις και λίγο μαθαίνουμε ότι μια ουσία έχει κάποιες ε, ε, δράσεις και επιπτώσεις που μέχρι χτες αγνοούσαμε. Δηλαδή πρέπει να είναι μια διαρκής ε, διαδικασία αυτή, όχι σε φάσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, Ράιντ και από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που ήρθατε και μας δώσατε όλη αυτή την ευρύτατη επισκόπηση της Προεδρίας σας. Ένα συγκεκριμένο θέμα θέλω να αναφέρω και να ακούσω την άποψή σας και τα σχέδιά σας. Ε, ε, αυτό το θέμα για τη στιμαριθμική αναπροσαρμογή των επιδομάτων τέκνων ε, ανάλογα με τη χώρα που ζουν τα παιδιά. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη αυτή η συζήτηση και γίνεται και στη Γερμανία αυτό τον καιρό, την πατρίδα μου. Οι Ευρωπαίοι τώρα έρχονται αντιμέτωποι ο ένα στον άλλον. Ένα αυτοματισμό, μια κοινωνία απέναντι στην άλλη. Υποδαβλίζονται διάφορα μίση και πάθη και στο Ηνωμένο Βασίλειο από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά η εκστρατεία για το δημοψήφισμα του Brexit με το αποτέλεσμα που είδαμε όλοι. Ήταν πάρα πολύ εχθρική η συζήτηση αυτή, αντιευρωπαϊκή, μα το θέμα είναι θεμέλιο ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεταχείριση ε, όλων των πολιτών ανεξαρτήτως προέλευσης ή καταγωγής. Και για μένα είναι σημαντικό να μάθω τι προτίθεται να κάνει η Ρουμανική Προεδρία για να αντικρούσει αυτή τη συζήτηση. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε αυτό να τρέχει και να εκπνεύσει. Το είδαμε στη Μεγάλη Βρετανία ε, και που κατέληξε. Σε κάποια κράτη-μέλη προχωρούν και σε νομοθετικές ρυθμίσεις για την αναπροσαρμογή των επιδομάτων τέκνων ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχεται ο εργαζόμενος ή ζουν τα παιδιά του. Γιατί αυτό θα καταλήξει ε, σε ε, καταστάσεις τελείως αντίθετες με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιφατικές μεταξύ τους. Έχετε σχέδια στρατηγική. Ευχαριστώ. Thank you. And the last... Ευχαριστώ και η τελευταία ερώτηση του κυρίου Κούκαν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Υπουργέ, καλωσορίσατε στην Επιτροπή Ευασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Είναι η πρώτη σας αυτή η ιστορική Ρουμανική Προεδρία και όλοι σας θυμίζουν ότι θα είναι δύσκολη, σημαντική, απαιτητική. Ισχύουν όλα αυτά. Και στην ίδια ανάσα όμως θα έλεγα ότι είναι και μια χρυσή ευκαιρία για σας να δείξετε πόσο καλοί είστε και να δείξετε τι αξίζεται. Κάντε το για να κλείσετε τα στόματα όλων αυτών που σας κατηγορούν ε, ε, ότι δεν μπορεί η Ρουμανική Προεδρία να είναι μια αποτελεσματική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλή σας τύχη. Θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα. Η δική σας συνεργασία με την Επιτροπή μας είναι κάτι το οποίο όλοι εκτιμούμε πάρα πολύ και θα εκτιμήσουμε στο μέλλον. Διάβασα με ενδιαφέρον το πρόγραμμα της Προεδρίας σας και εστιάζεται στην κινητικότητα των εργαζομένων που είναι ένα θέμα πάρα πολύ ακαθόδες και επίμαχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά είναι ταυτόχρονα και στη βάση των τεσσάρων ελευθεριών μας. Υπό την έννοια αυτή έχω μια πολύ σύντομη και μικρή ερώτηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αρχή ε, ε, Εργασίας, η Την αναφέρατε εισαγωγικά. Ε, εξ όσων έχω καταλάβει, η δική σας Προεδρία θέλει να καταλήξει σε συμφωνία για την ίδρυση αυτού του νέου οργανισμού, Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Και στις προγραμματικές σας δηλώσεις λέτε και παραθέτω μαζί με τα κράτη-μέλη η Ρουμανική Προεδρία θα διερευνήσει τι καλύτερε δυνατότητε για να ορίσουμε το ρόλο και τι ευθύνε τη μελλοντική αυτή αρχή και ε, στοχεύουμε να ολοκληρώσουμε ε, τις ε, διαπραγματεύσεις για αυτό το θέμα. έξι της παράθεσης. Σίγουρα μπορεί να βελτιώσει την κινητικότητα των εργαζομένων για τους μετακινούμενους εργαζόμενους και εταιρείε. Παρ' όλα αυτά, θα θέλαμε να μάθουμε πώς προτίθεται η Προεδρία σας να αντιμετωπίσει το θέμα της επιλογής της έδρας. Ιδιαίτερα, πότε θα το κάνετε αυτό. Γιατί ενδιαφέρεται η Σλοβακία. Ελπίζω να ερμηνεύσατε σωστά για ποιο λόγο σας κάνω αυτή την ερώτηση. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέμβασή σας, λέει η Πρόεδρος, και θα δώσω το λόγο στον Υπουργό για να απαντήσει. Ακούσατε τι είπαν οι βουλευτές έχουν αποθέσει μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες στη Ρουμανική Προεδρία και πολλή δουλειά έχετε και λίγο χρόνο. Σας δίνω ξανά το λόγο, Υπουργέ, για να προσπαθήσετε να απαντήσετε. Ε, περιμένουμε πολλά από εσάς, παρακαλώ. Mulțumesc, doamnă președintă. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους βουλευτές, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για τις ερωτήσεις που μου έχουν απευθύνει. Κράτησα σημειώσει ε, λίγο ανάκατα. Ελπίζω να καταφέρω να βγάλω μια άκρη και να είμαι σε θέση να σε απαντήσω με ικανοποιητικό τρόπο. Αν δεν τα καταφέρω, παρακαλώ να επανέλθετε και να ε, ξαναπροσπαθήσω στη συνέχεια. Μην διστάσετε λοιπόν. Γιατί είναι πολύ σημαντικοί οι προβληματισμοί που μα διακατέχουν ε, όταν καθορίζουμε το χρονοδιάγραμμα εργασιών τη Ρουμανική προεδρία. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα χρονοδιάγραμμα όσο δυνατόν πιο πλήρε, πιο εμπεριστατωμένο, για να κάνουμε τα πράγματα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τρόπο και για να βοηθήσουμε όσο δεν το περισσότερο μπορούμε, όσο το περισσότερο μπορούμε, για να ε, καρπίσει η προεδρία, η μας και να φέρει αποτελέσματα. Έχω την εντύπωση λοιπόν, και αν δεν απατώμε, ε, ότι ξεκίνησα την παρουσίασή μου λέγοντας κάτι που χρειάζεται και τώρα να επαναλάβω. Είπα στην αρχή της παρέμβασής μου για εμάς το ότι έχουμε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αποδείξουμε σε ποιο βαθμό υπερασπιζόμαστε και προάγουμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το εννοώ το λέω σοβαρά, σοβαρότατα. Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να παγιώσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα κοινωνικής ολοκλήρωσης, για να αναδείξουμε και να θωρακίσουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Και νιώθω ευγνωμοσύνη, διότι ε, βλέπω μέσα από τις διάφορες ερωτήσεις σας ότι ε, τελικά... Ε, μας διαβιβάζετε τις βασικές ανησυχίες της δικές σας και των Ευρωπαίων πολιτών και παρόλο που έχουμε λίγο χρόνο αυτό σημαίνει ότι θα μας βοηθήσετε για να ολοκληρώσουμε την εξέταση των φακέλων με όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικό τρόπο προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Κύριε Κάσα, Στρέφομαι σε εσά για να σας πω το εξή. Όταν παρουσιάσαμε τις προτεραιότητες τη Ρωμανικής προεδρία, ήδη είπα ότι η συμφιλίωση μεταξύ ε, επαγγελματική και οικογενειακή προσωπικής ζωής αποτελεί ε, μία από τις προτεραιότητές μας. Θα δώσουμε λύσει που θα επιτρέψουν σε όλους τους εργαζόμενους να έχουν ίσα δικαιώματα και θα προσπαθήσουμε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για αυτό το θέμα τη συμφιλίωση οικογενειακή και επαγγελματική ζωή. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό ε, Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση και το φάκελο το σχετικό. Έχω την τύχη να μπορώ να βασίζομαι σε εξαιρετικού διαπραγματεύτέ και εδώ στι Βρυξέλλες αλλά και στη Ρουμανία στο Υπουργείο μου. Επομένω, στο Συμβούλιο προσπαθούμε να καταλήξουμε, να φτάσουμε σε αποτελέσματα το συντομότερο δυνατόν. Και θα ήθελα εδώ να ανοίξω μια παρένθεση για να πω το εξής. Από το 1995 εργάζομαι στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης της χώρας μου. Και γιατί το λέω αυτό. Διότι προσωπικά εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά το θέμα των δικαιωμάτων, των ελευθεριών, των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Είναι πράγματα που γνωρίζω πολύ καλά. Όλα τα δικαιώματα που εκπορεύονται από τον κοινωνικό πυλώνα. Δεν μου είναι κανένα άγνωστο. Κλείνω λοιπόν την παρένθεση εδώ, ε, την προσωπική, για να σας μιλήσω για την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας ε, στον στο να, κατα... Ε, να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις σε αυτό το σκοπό αυτός μας απασχολεί κυρίως. Στην πλειονότητα των θεμάτων συμπίπτουν οι απόψει των δύο θεσμικών οργάνων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Πρέπει να δούμε ποια θα είναι η πιο ταχεία διαδικασία για τη λήψη απόφασης χωρίς αυτό να επηρεάσει ε, την ε, χρονική διάρκεια για την έγκριση κατά τη διάρκεια της παρουσίας θητείας. Δηλαδή πρώτα ε, πρέπει να διαπραγματευτούμε για την νομοθετική πράξη και μετά τα υπόλοιπα. Από εκεί και πέρα, ό,τι αποφασιστεί στους τριμερείς διαλόγους, θα ε, το αξιοποιήσουμε, θα στηριχθούμε πάνω σε αυτό για να πετύχουμε προστιθέμενη αξία. Όποιο και να είναι το θέμα της διαπραγμάτευσης ε, και του εκάστοτε τριμερούς διαλόγου. Επομένως, επαφίεμαι στους συνεργάτες μου, σε εσάς που δουλεύουν εδώ στις Βρυξέλλες. Κάποιοι από εσά μας είπατε ότι είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι. Τι να κάνουμε. Αφού έχουμε τόσο λίγο χρόνο, πρέπει να προσπαθήσουμε για το μέγιστο. Και πρέπει να συνεργαστούμε με εσάς. Βασίζομαι λοιπόν στη βοήθειά σας. Θεωρώ και εκτιμώ ότι θα μας βοηθήσετε για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Να ολοκληρωθεί η εξέταση διαφόρων φακέλων κοινωνικών υποθέσεων που είναι τόσο σημαντική για τον Ευρωπαίο πολίτη. Για παράδειγμα, ε, τα επιδόματα για το όταν έχει κανείς ανηλίκους στον οικοκυριό του και τον βαρύνων. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ενιαία αγορά με σαφείς αρχές, ε, ορθές αρχές και να ε, ε εποφελούνται όλα τα κρατημέλη. Θέλουμε να στηριχθεί η ισχύουσα νομοθεσία, η κείμενη νομοθεσία. Και κάθε φορά που υπάρχει η παραβίαση, η καταστρατήγηση αυτών των αρχών, η παράβαση, ε, θεωρούμε ότι υπάρχουν ε, μηχανισμοί και ανάλυσης της κατάστασης και κύρωσης ε, για τις αστοχίες αυτές και τις παρατυπίες. Κυρία Λάμπερτ, μου θέσατε ερώτημα για την κινητικότητα των εργαζομένων. Και έχω να σας πω ότι αναζητούμε συγκεκριμένες λύσεις, απτές, πρακτικές θα έλεγα. Για τον κανονισμό 883, εκεί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που διευκολύνουν τη διαδικασία για την κινητικότητα των εργαζομένων. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να σημειώσουμε κάθε δυνατή πρόοδο, ωστόσο είναι αληθές ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες. Προσπαθώ ακόμα να ξεκαθαρίζω τις σημειώσεις μου που πήρα εντάχει ε, καθώς ο χρόνων εσείς ε, διατυπώνατε τις ερωτήσεις σας. Ναι, έρχομαι τώρα στον κύριο Πάβελ και στα εθνικά μέτρα ρώτησε κάτι για αυτό το θέμα. Και έχετε δίκιο κύριε, ε, κύριε Πάβελ. Έχουμε 4 εκατομμύρια Ρουμάνους πολίτε οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τη Ρουμανία, Ρουμανία, δουλεύουν αλλού και δεν φέρνουν, δεν κομίζουν καμία προστιθέμενη αξία στη δική μου χώρα. Και γι' αυτό η κυβέρνησή μου και η Πρωθυπουργό σε στενή συνεργασία με τι συνδικαλιστικέ οργανώσει, αλλά και με την εργοδοσία, τι εργοδοτικέ οργανώσει, έχουν έρθει σε επαφή με του εκπροσώπους τη Ρουμανική ομογένειας στο εξωτερικό για να υπάρξει ένα πρόγραμμα υποτροφιών για την επιστροφή των εργαζομένων έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες εργασιακό δυναμικό που έχουμε. Δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες γιατί είναι εθνικό θέμα ενώ είναι κοινοβουλευτική η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, η κοινωνική Ευρώπη είναι κάτι που μας ενδιαφέρει και ως Ρουμανική Προεδρία θέλουμε ο Ευρωπαίος πολίτης να είναι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της Ρουμανικής Προεδρίας, της δικής μας Προεδρίας κάθε προεδρία πρέπει να ε, λειτουργεί ε, έτσι ώστε να ανεβαίνει το βιωτικό επίπεδο των Ευρωπαίων πολιτών και για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να συνεργαστούμε με εσάς. Ε, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι άλλο ένα πρόβλημα και άλλη μια προτεραιότητα για μας όπως έχουμε ήδη πει. 5,2% είναι το σχετικό νούμερο για τη Ρουμανία ενώ 16% είναι κατά μέσο όρο το μισθολογικό χάσμα στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά μέσο όρο πάντοτε. Η κυβέρνηση λοιπόν έχει προδρομολογήσει ένα πρόγραμμα πρόσβαση σε πόρους για τη δημιουργία ε, νεοφιών επιχειρήσεων. Startup Nation λέγεται το πρόγραμμα αυτό. Το 50% αυτών που έχουν λάβει ενισχύσεις είναι γυναίκες. Και εμεί στην Ρουμανία είναι κάτι που μα ενδιαφέρει ιδιαίτερω και είναι κάτι το οποίο προσέχουμε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία, την εμπειρία που έχουμε αθροίσει, που έχουμε συσσωρεύσει και να την ε, αξιοποιήσουμε ή να τη χρησιμοποιήσουμε σε όλε τι συζητήσει και του τριμερεί διαλόγου στου οποίου προεδρεύουμε και θα προεδρεύσουμε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, Εάν κάποιος από τους παριστάμενους θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να μας ζητήσει βοήθεια ή θέλει να μας καλέσει ή να το καλέσουμε σε οποιαδήποτε συνέδριο που οργανώνει ο ίδιος ή οργανώνουμε εμείς, ε, πρέπει να το πράξει. Είναι ευπρόσδεκτος. Σε κάθε περίπτωση θα προωθήσουμε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για το θέμα αυτό, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, ε, για τον καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος και των λοιπόν ανισοτήτων που επικρατούν στην αγορά εργασίας μεταξύ ε, των δύο φύλων. Για τι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας, να σας πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μας, η υγεία του Ευρωπαίου πολίτη όταν εργάζεται. Η οδηγία για τις καρκινογόνες και μεταλλαξιογόνες ουσίες είναι ένας πολύ καλός τρόπος να βελτιώσουμε την υγεία των εργαζομένων στο φόρο εργασίας. Και ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις για αυτή την οδηγία θα ολοκληρωθούν κατά τη διάρκεια της δικής μας προεδρίας. Ελπίζω λοιπόν ότι κατάφερα να απαντήσω στις ερωτήσεις σας και ελπίζω ότι κατάφερα να σας παραθέσω τους στόχους μας τους οποίους θα πετύχουμε μόνο με τη δική σας βοήθεια. Αν τώρα κάτι μου έχει ξεφύγει, αν σε κάτι δεν έχω απαντήσει λεπτομερώς και επαρκώς, παρακαλώ ε, να επανέλθετε. Να ξέρετε όμως ότι έχετε την πλήρη στήριξή μας, τη δική μου προσωπικά και αυτή των βοηθών και συνεργατών μου, τους οποίους ευχαριστώ, δημόσια εδώ. Ευχαριστώ και εσά και θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια όλου του συναδέλφου από τα Ρουμανικά Υπουργεία και από τη μόνιμη Ρουμανική Αντιπροσωπεία για αυτή την κοινή συλλογική μα προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Uh, ε, προσπαθήσατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Μας είπατε ότι έχετε τη φιλοδοξία να ολοκληρώσουμε όσο γίνεται περισσότερα νομοθετήματα από όσα εκκρεμούν πριν φτάσουμε στην προεκλογική περίοδο και μπούμε στην προεκλογική εκστρατεία. Δηλώσατε πρόθυμος να συνεργαστείτε μαζί μας, να απαντάτε σε τυχόν ερωτήσεις που θα έχουμε. Θα παραμείνουμε σε επαφή και σε πολύ στενή επικοινωνία. Και προσβλέπουμε πάρα πολύ σε όλους τους τριμερείς διαλόγους στους οποίους θα συναντηθούμε ξανά για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να δώσουμε και αποτελέσματα στους Ευρωπαίους πολίτες. Ειδικά επειδή μας περιμένουν και εκλογές. Uh, σας ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας και είστε πάντα πρόσδεκτος. Ευχαριστώ πολύ. Ε, σας παρακαλώ μια στιγμή, ε, ήθελα κάτι να προσθέσω που ξέχασα. Να απαντήσω σε μια ερώτηση για το, τη δέσμη σχετικά με την κινητικότητα. Φυσικά και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το σύνολο των νομοθετημάτων, αλλά θα πρέπει να συνενεθούμε και με τους συναδέλφους μας του Υπουργείου Μεταφορών, γιατί εκεί βρίσκονται τα μεγαλύτερα προβλήματα. Ε, συνεργαζόμαστε πάντως για να δούμε από κοινού αυτά τα θέματα. Thank you also, Mr. Ευχαριστώ και σας κύριε Σόγκορ για την απάντηση και σας ευχαριστώ και ο κύριο Σόγκορ που απαντήσατε ε, στην ερώτησή του. Στο καλό να πάτε και να μας ξανάρθετε. our voting session, but we'll, uh, we will uh, start at 4 o'clock so that all members can be here. Περιμένουμε να ξαναρχίσουμε στις 4. Έχουμε ένα διαλυματάκι 9 λεπτών. And then we'll start uh, at uh, 4 o'clock sharp. Thank you very much. Υπότιτλοι

Okay, then we start the voting session and Ας αρχίσουμε λοιπόν, ε, φίλοι μου, τις ψηφοφορίες. Έχουμε πρώτα την ε, απαλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή του Γενικού Προϋπολογισμού της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχίζουμε με την παράγραφο 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7α υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 2 ψηφίζεται τέλος της ψηφοφορίας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 Και τώρα πρέπει να ψηφίσουμε με ονομαστική κλίση για το σχέδιο χρωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται. Τέλος της ψηφοφορίας. 40 υπέρ, 2 κατά και μια αποχή. Ευχαριστώ. Την κυρία Χάρκιν, την αστυγητρία. Δεύτερο σχέδιο χνομοδότησης, κυρία Χάρκινγκ. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη Επαγγελματική Κατάρτιση, ΕΝΤΕΦΟΠ, Συμβαστική 1, υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ελέγχουμε την τροπολογία 2. Άρχεται. Τέλος. Εγκρίνεται. 24 ψήφοι υπέρ, 19 κατά. Τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε την τροπολογία 6 τέλος με προφορική τροπολογία ναι εγκρίνεται με 30 ψήφους υπέρ 12 κατά και 2 α, αποχές Παράγραφος 8β. Άρχεται. Τι ψηφίζουμε παρακαλώ. Ψηφίζουμε την παράγραφο 8β, τροπολογία 7. Α, μάλιστα, εντάξει. Μπορείτε απλά να σηκώσετε τα χέρια σας αν θέλετε, είναι πιο απλό. Ποιοι είστε υπέρ. Για περιμένετε. και Εγκρίνετε. Τώρα, ονομαστική κλίση για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία, τέλος της ψηφοφορίας, εγκρίνεται με 39 ψήφους υπέρ, 3 κατά και 2 αποχές. Τώρα, απαλλαγή όσον αφορά την εφαρμογή του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού ιδρύματο ε, για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωση και εργασία στο Eurofound. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 είναι μια προφορική τροπολογία. Για την 9. Τροπολογία είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε για το σχέδιο γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση. Τέλος της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται με 43 ψήφους 42 ε, υπέρ, συγγνώμη, μία κατά και δύο αποχές. Πάμε στο σχέδιο γνωμοδότησης για το όσα γράφος 2, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3, υπέρ, κατά, ελέγχουμε. Τροπολογία 3. Άρχεται. Και τέλος ψηφοφορίας. Ένας παραπάνω είστε στο ΕΛΚ. Μάλιστα, 25 υπέρ, 20 κατά. Άρα εγκρίνεται. Προχωράμε στην τροπολογία 4. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 5 τροπολογία 9. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία εδώ έχει αποσυρθεί και προχωράμε στην τροπολογία 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7, τροπολογία Μάλλον έχει καταπέσει, συγγνώμη. Πάμε στην παράγραφο 8, τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. ε, παράγραφος 9, τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Ε, ε, ε, ναι, με συγχωρείτε. Ε, απορρίπτεται, ήθελα να πω. Then we go to the roll call vote to the end. Ονομαστική κλίση για την γνωμοδότηση όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται τέλος, εγκρίνεται με 42 ψήφους υπέρ, 2 κατά και μία αποχή. Και σας ευχαριστώ. Προχωρούμε. Απαλλαγή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ETF. Παράγραφος 1. Ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 1. Ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τι έχουμε εδώ τώρα. Πάμε μέσω στην τελική ψηφοφορία που αρχίζει τώρα και τελειώνει ευθύ αμέσω. 42 ψηφίπερ 2 κατά και 2 εποχές. Ευχαριστούμε λοιπόν τον συγητή και προχωρούμε στο σχέδιο γνωμοδότησης για την απαλλαγή ε, του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Οργανισμών για το οικονομικό έτος 2017 έλεγχος επιδόσεις ε, και ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 1 ήταν αυτή η τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 4 ψηφί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το σχέδιο της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε, η ονομαστική είναι η ψηφοφορία όπως ε, πάντα. Αρχίζει τώρα. Πέρας. 42 ψήφισαν υπέρ, ένας κατά και δύο απήχαν. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες. Την άλλη φορά θα είμαι καλύτερα έτσι από φωνή και γενικότερα. Για να μπορέσω να κάνω πιο γρήγορα τις ψηφοφορίες. Yeah. Ξέρετε ότι έχουμε και άλλο θέμα όλοι φυσικά στην ημερησία διάταξη. Έχουμε ακόμα ένα θέμα. Ε, μια παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα μας ενημερώσει. Great Για πολύ σημαντικά για μας θέματα. Κατ' εξοδότηση κανονισμός της Επιτροπής είναι το θέμα μας. και με χαρά θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θέλω και να μείνετε και να ακούσετε. Θα χαρώ πολύ. Έχετε παρακαλώ το λόγο. Ελάτε εδώ παρακαλώ, εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank Σας ευχαριστώ που ήρθατε και σας δίνω μέσα στο λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλα τα αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Θα ήθελα λίγο να σας παρουσιάσω ε, την ε, παρουσίαση μου στα άρθρα 14.1 του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εξουσία ε, να ε, προχωρεί σε κατεξοδότηση ε, κανονισμούς για την απλούστευση των πληρωμών και των σχετικών κλιμακίων. Αυτό εγκρίθηκε το 2015 και συνεχώς αναπροσαρμόζεται, ανανεώνεται γιατί καταθέτουν συνέχεια προτάσεις τα κράτη-μέλη. Πού βρισκόμαστε ε, με τις τροποποιήσεις, πόσες τροποποιήσεις έχουν γίνει, ε, ποια είναι τα κόστη που καλύπτονται από αυτές τις απλουστευμένες διαδικασίες. Πρώτα, το άρθρο 14.1 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρεί ε, ε, σε κατεξουδότηση πράξης για το απλοποιημένο κόστος και αυτό μπορεί να ισχύει για οποιοδήποτε κράτος μέλος και για κάθε είδους πληρωμή. Μέχρι τώρα ε, έχουμε εγκρίνει κατά αποκοπή ποσά μετά από αίτημα των κρατών μελών με συγκεκριμένα δεδομένα, στοιχεία, στατιστικές και μεθόδους που έχουμε συμφωνήσει από κοινού Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Η διαδικασία αυτή δίνει πολύ μεγάλη νομική βεβαιότητα στα κράτη-μέλη και τις διαχειριστικές αρχές, βελτιώνει και τις λογιστικές πρακτικές γιατί τις ευθυγραμμίζει. Ε, πρακτικές λογιστικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών. Και ε, με τη σειρά του αυτό καλύπτει και πολλά περισσότερα έξοδα, περισσότερα είδη δαπανών βάσει υπολογισμών που έχουν κάνει προτάσεις του στα κράτη-μέλη. Υπήρξε και μια ομάδα υψηλού επίπεδου πριν από λίγα χρόνια που ενέκρινε κάποια κριτήρια και κατέληξαν ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη απλούστευση για το κόστο. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναπτύξουν αυτά τα κλιμάκια και τις δυνατότητε, με όλες τις αντιστοιχές, τα δεδομένα και τα στοιχεία που διαθέτουν. Και επίσης ήδη έχουμε αναπτύξει μια διαδικασία πλουσεμένου κόστου σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στοιχεία της Eurostat αλλά και πολλέ ε, μελέτες και εκθέσει. Και με το νέο κανονισμό καλύπτουμε άλλα τρία είδη ε, δαπανών και πληρωμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι πολύ μεγάλη και η πολιτική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, γίνει γενική πρακτική αυτή η απλουστευμένη διαδικασία με στόχο να καλύπτουμε περίπου τις μισές δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο. Να καλύπτονται δηλαδή από αυτή την απλοποιημένη διαδικασία. Ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι προχωρούμε καλά. Στην ε, τρέχουσα τροποποίηση που είναι η έκτη υπάρχουν διάφορα κράτη-μέλη που προτείνουν απλουστευμένες διαδικασίες και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προτείνει άλλες τρεις. Θα μπω σε λεπτομέρειες στις επόμενες διαφάνειες. Ο κατεξοδότης κανονισμός είναι πάρα πολύ μικρός. Ξέρετε ότι έχει μόνο τέσσερα άρθρα αλλά η ουσία του κανονισμού είναι στα παραρτήματά του. Έχουμε ένα παράρτημα ανακράτος μέλος και όταν έρχεται το κράτος μέλος με μια νέα πρόταση, προστίθεται η πρόταση αυτή στο παράρτημα. Αν θέλουν να το τροποποιήσουν για να αλλάξουν τα δεδομένα και τα στοιχεία, παραμένουν στο ίδιο παράρτημα. Περιλαμβάνει το παράρτημα ε, τον ορισμό των δικτών, τις μονάδες μέτρησης και τις προτάσεις ε, των κρατών μελών και επίση, όταν το ζητούν τα κράτη-μέλη μπορούν και να προσαρμόζονται τα ποσά ανάλογα με τα νέα οικονομικά δεδομένα. Ε, πώς έχει μέχρι τώρα η κατάσταση. Ο κανονισμός εγκρίθηκε αρκετό καιρό τώρα, το 2015. Πέντε φορές έχει τροποποιηθεί, καλύπτει 18 κράτη-μέλη και ε, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια προστευμένη διαδικασία τέτοιο κλιμάκιο για την παιδεία. Και με τον τρέχοντα κανονισμό, όπως τροποποιείται τώρα, με την έκτη τροποποίηση, θα έχουμε περίπου 10 δισεκατομμύρια ε, των δαπανών του ESF που θα μπορούν να πιστοποιούνται με την απλουστευμένη αυτή διαδικασία. Και η έκτη τροποποίηση αφορά 18 κρατη είναι ένα που έχει ε, προσθεθεί ε, σύνολο 19 γιατί η Βουλγαρία πρότεινε μια τέτοια απλοποιημένη διαδικασία ε, για την επαγγελματική κατάρτιση και την εκπαίδευση. Ε, τροποποιούμε λοιπόν τα παραρτήματα για τη Γαλλία, Τσεχία, Σλοβακία, Αυστρία, Ρουμανία, Κύπρο και Κροατία και προτείνουμε το τυποποιημένο κλιμάκιο μοναδίου κόστους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, κατάρτιση ανέργων, τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών και για στοχευμένες δράσεις. Ε, βλέπετε εδώ γιατί για τη Βουλγαρία, για μοναδίο κόστος εκπαίδευσης βάση αποτελεσμάτων. Στη Γαλλία χρειάστηκε διευκρίνηση της ορολογίας. Η τσεχική δημοκρατία είναι ηγέτη σε αυτή την προσπάθεια. Μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί 32 τυποποιημένα κλιμάκια μοναδίου κόστους. Και τώρα περιμένουμε την 7η τροποποίηση όπου προτείνει η τσεχική δημοκρατία επιπλέον απλοποίηση γιατί πραγματικά τότε θα αποδειχτεί πρωταθλητής ε, σε αυτή τη διαδικασία όταν στέλνει ε, αποδείξεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, πληρωμές. Στη Σλοβακία ε, χρησιμοποιείται για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην Αυστρία. Έγιναν κάποιες διευκρινήσεις για το μισθολογικό κόστος, για τη δημοτική εκπαίδευση, για την εκτουσύνεγγης παροχή συμβουλών και ε, τη διαχείριση υπηρεσιών επαλήθευσης και τις ε, αμοιβέ. Για την ε, Ρουμανία έχουμε ε, δύο κλίμακες με δύο κόστους. Για την επαγγελματική κατάρτιση και το δεύτερο είναι για την ε, ανεργία και τα επιδόματα ανεργίας. Μάλλον για την βοήθεια για την απασχόληση. Και με την Κύπρο πάλι αντίστοιχα για κατάρτιση και επαγγελματική εκπαίδευση και για την Κροατία νέο μοναδιακόστος κόστο που έρχεται να προσθεθεί στο προηγούμενο ε, επαγγελματική κατάρτιση, βοήθεια για την απασχόληση και μηνιαία αποζημίωση για τα οδηπορικά των συμμετεχόντων. Όλα αυτά ε, που εγκρίθηκαν με την πέμπτη τροποποίηση ε, έχουν αλλάξει για να καλύψουμε και την Ελλάδα που τώρα συμμετέχει, γιατί όταν έγινε η πέμπτη τροποποίηση δεν είχαμε αρκετά στοιχεία, τώρα έχει ενταχθεί και η Ελλάδα σε αυτό το πρόγραμμα και μετά από κάποια αιτήματα των κρατών μελών διευκρινίσαμε το πώς θα αντιμετωπίζουμε ε, τα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης μερικού χρόνου όμως, όχι πλήρους ωραρίου. Τώρα υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία ενιαία που μπορούν να χρησιμοποιούν όλα τα κράτη-μέλη και όλες οι διαχειριστικές αρχές έτοιμο παράδοτη, ε, γιατί αυτό είχε ζητήσει και η ομάδα υψηλού επίπεδου, να υπάρχουν πολλέ περισσότερες επιλογές ε, σε ό,τι αφορά τις τυποποιημένες κλίμακες μοναδιαίου κόστους. Ε, πήρε βέβαια λίγο χρόνο για να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία, όλα τα δεδομένα, από βάσεις δεδομένων, από πληροφορίε που είχαμε για την αγορά εργασία. Ε, τα επιχειρηματικά μοντέλα, τρόπος που προκυρήσονται οι διαγωνισμοί, οι προμήθειες κτλ. για να καταλήξουμε σε ένα πανευρωπαϊκό επίπεδο και το κόστος να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές δαπάνες και τις καταβληθήσεις ε, για διάφορες μορφές ε, κατάρτισης και επαγγελματική εκπαίδευσης. Τρεις είναι οι τομείς λοιπόν στη νέα πανευρωπαϊκή κλίμακα, ε, κατάρτιση ανέργων, υπηρεσίες παροχής συμβουλών και κατάρτιση εργαζομένων. Έχουμε και πιο ε, περιφερειακή διάσταση στην εφαρμογή για τα κράτη-μέλη όταν υπάρχουν ε, περιφερειακές διαφορές ως προς το κόστος για χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Βασίζεται αυτό σε στοιχεία και δεδομένα της Eurostat σχετικά με τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες μίας χώρας δεν επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να επιλέγουν τι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις απλουστοδευμένες διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τις εθνικές. Αυτό δεν γίνεται δεκτό. Ε, δεχόμαστε μόνο την ευρωπαϊκή διαδικασία και όχι την εθνική που να βασίζεται σε δικά τους εθνικά στοιχεία. Για ποιο λόγο, γιατί έτσι εκτιμούμε καλύτερα το κόστος. Έχουμε... Έχουμε πολλέ πληροφορίε σε εθνικό επίπεδο. σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι λιγότερε και λιγότερο συγκρίσιμες. Τα κράτη-μέλη λοιπόν γνωρίζουν καλύτερα ε, το κόστο και τι συνθήκε που επικρατούν και τα στοιχεία και μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ευρωπαϊκή διαδικασία, ε, ακόμα και για νέες χρήσεις που μπορούν να προταθούν και να είναι επιλέξιμες για τη διαδικασία αυτή. Τώρα θέλω να σα ενημερώσω ότι εργαζόμαστε αυτό το καιρό για την 7η τροποποίηση του κανονισμού αυτού, του κατεξοδότηση και θα εγκριθεί περί τα μέσα Φεβρουαρίου και νωρίτερα. Υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη που περιμένουν να εγκριθεί αυτή η τροποποίηση για τους δικούς τους εθνικούς λόγους και ελπίζω να έχω την ευκαιρία να ξανάρθω ε, προσεχώς αμέσως μετά τα μέσα Φεβρουαρίου για την 7η τροποποίηση. Αν δεν υπάρξει καμία αντίρρηση για να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν αυτό το πολύτιμο εργαλείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Είναι λίγα τα μέλη στην αίθουσα, όμως ε, όσοι είναι εδώ θέλουν να πάρουν το λόγο. Ε, χρειάζεστε κάποια διευκρίνηση, κύριε Ντέτσιεν. Κύριε Πυρίνσκι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, να σας καλωσορίσω, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσίαση, γιατί ασχολείται με ένα ζήτημα που έχει συζητηθεί τα μάλα, πώς δηλαδή χρησιμοποιεί κανείς την απλουστευμένη επιλογή κόστους και πώς μπορεί να τη διαδώσει, να χρησιμοποιηθεί αυτή η επιλογή πιο ευρέως και να αξιοποιηθεί περισσότερο. Γιατί αυτό είναι σημαντικό για τη χρηστή οικονομική διαχείριση και για την αποτελεσματική αξιοποίηση και χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θα ήθελα παρόλο που από τα λεγόμενά σας θεωρώ ότι προκύπτει. Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να ρωτήσω το εξής γιατί ξέρουμε ότι σε ορισμένε περιπτώσει τα κράτη-μέλη, κάποια κράτη-μέλη ήταν διστακτικά. Δίσταζαν να προσφύγουν σε αυτή την επιλογή απλουστευμένου κόστου για διάφορου λόγου. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε τις διάφορες δυσκολίες, σας έχουν γίνει παρουσιάσεις για τα εμπόδια, για τις δυσκολίες. Πιστεύω ότι έχετε υπογραμμίσει ότι είναι κάτι το οποίο σας έχει προβληματίσει και ε, ξέρετε πώς να το ξεπεράσετε. Μπορείτε να μας αναπτύξετε αυτό το θέμα, ποιες είναι οι απαντήσεις που θα δώσετε ε, για να πείσετε, για να αξιοποιηθεί περισσότερο αυτή η ευκαιρία η οποία έχει πολλές δυνατότητες και θα μπορούσε να αποβεί πολύ χρήσιμη και για τα κρατημέλη αλλά και για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα Στη συζήτηση για το ευρωπαϊκό επίπεδο είπατε ότι βασιστήκατε στα δεδομένα και τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat καθώς και τις έρευνες που έχει αυτή διεξάγει. Να σας αναφέρω κάτι που συνέβη σήμερα το πρωί. Η κυρία Ουσκόπη, πρόεδρος, είχε ασχοληθεί ε, για την οριστικοποίηση ενός τριμερούς διαλόγου με το Συμβούλιο και ε, για τον κανονισμό για τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για τις έρευνες κοινωνικών θεμάτων, κοινωνικής θεματολογίας για τις κοινωνικές στατιστικές. Και ένα από τα τελευταία ζητήματα που είχαν μείνει και που επρόκειτο να συζητηθούν ήταν το εξή. Σε ποιο βαθμό οι υπηρεσίες, οι οργανισμοί, οι αρχές μέσα στο Ευρωπαϊκό Σύστημα θα τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούν δεδομένα δεδομένα από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες και σε ποιο βαθμό θα είναι σε θέση να συμφωνήσουν ότι θα μπορούσε η Eurostat να καλεί τις υπηρεσίες όταν αναπτύσσει και βελτιώνει ε, τα συστήματά της και τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας να καλεί τις ευρωπαϊκές αρχές και υπηρεσίες. Και αυτό θα ήταν ενδιαφέρον. Δηλαδή η Επιτροπή θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει με το δικό σας προσωπικό και τελικά να δείτε σε ποια σημεία εντοπίζεται μια χρήσιμη συνεισφορά. Ε, δηλαδή, μια βελτιωμένη Eurostat και βελτιωμένα αποτελέσματα της Eurostat σε ποια σημεία θα μπορούσε αυτό να είναι εξαιρετικά βοηθητικό, για ποια θέματα. Αλλά έχει σημασία και με τις ε, υπηρεσίες που εγκρινούν τους προϋπολογισμούς. Έχουμε συνεδρίαση ψηφοφορίας για το 2017 και νομίζω ότι έχουμε αρκετή αξιοπιστία γιατί εγκρίναμε τους προϋπολογισμούς των διαφόρων οργανισμών με ε, απρόσκοπτο τρόπο. Επομένως, αυτό που μας παρουσιάσατε σήμερα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, αποφασιστικότητά σας και θέλω να εκφράσω την ετοιμότητά μας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Η ομιλήτρια παρακαλώ, η κυρία Σούκοβα. Ευχαριστώ κύριε Πυρίνσκι. Θα μπορούσα να ε, σχολιάσω επί μακρόν τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε αλληλεπίδραση με τα κράτη-μέλη και το πώς τα ενθαρρύνουμε. Έχουμε ένα δίκτυο διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστικών αρχών, ειδικά σε θέματα απλούστευσης και αυτό ήταν μια σταθερή προσπάθεια που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα τελευταία 4-5 χρόνια στο πλαίσιο της παρούσας ε, προγραμματικής περίοδου. Προσπαθούμε λοιπόν να εξηγούμε στα κράτη-μέλη και να αποδείξουμε ότι κάθε φορά που ισχύει και εφαρμόζεται η απλούστευση απλουστευμένη επιλογή κόστου στο ε, σύστημα πληρωμών. Δεν έχουμε συχνότητα σφάλματο που να εντοπίζεται από του ελεγκτέ. Δεν έχουμε ποσοστό σφάλματος. Οι ίδιες επιλογές για το προσεμένο κόστος μπορεί να ισχύσουν και στις σχέσεις μεταξύ κράτους μέλους διαχειριστικής αρχής και δικαιούχου και έτσι η, τα, όλη η δουλειά και όλες οι προσπάθειες εστιάζονται στα αποτελέσματα και όχι στα συστήματα λογοδοσίας και υπολογισμού και λογιστικών εγγραφών. Έχουν συζητηθεί οι τροπολογίες των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση με την ε, τεχνική μας ομάδα, ε, με τους τεχνικούς και όλες οι διαχειριστικές αρχές συμμετέχουν εκεί και εκπροσωπούνται. Είναι πολύ σημαντικό να το εξακριβώνουμε με τη διαχειριστική αρχή κάθε φορά ότι η μοναδιαία ε, τιμή ε, ε, αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα στα κράτη-μέλη. Τώρα, σε σχέση με την Eurostat, βεβαίω συνεργαζόμαστε στενά. Έχουμε τον ίδιο επίτροπο, έχουμε service level agreement, έχουμε συμφωνία σε επίπεδο τεχνικό των στελεχών μεταξύ υπηρεσιών. Ενίοτε υπάρχουν καθυστερήσεις, σημειώνονται καθυστερήσεις και εμείς κάθε φορά που δεν υπάρχουν στοιχεία έχουμε την ευθύνη και την υποχρέωση να επανεξετάσουμε και να επαναξιολογήσουμε την απλουστευμένη επιλογή κόστου εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία τη Eurostat για το εκάστοτε θέμα, έτσι ώστε ε, να, τα νούμερα να αντιποκρίνονται όσο να το περισσότερο στην πραγματικότητα όσο περισσότερη πληροφόρηση και καλύτερη πληροφόρηση δίδεται από τις Εθνικές Στατιστικές Αρχές στη Eurostat, τόσο πιο εύκολο είναι και για μας να αξιοποιούμε αυτά τα στοιχεία και να βασίζουμε τα συμπεράσματά μας σε αυτά τα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση η συνεργασία μας με την Eurostat είναι και θα παραμείνει πολύ στενή. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Εάν όχι, τότε να πω ότι η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι η 25η Ιανουαρίου και η καταληκτική προθεσμία για να γύρουν αντιρρήσεις στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και να ζητήσουν την παράταση της προθεσμίας είναι η 19η Μαΐου. Δεν έχει τελειώσει ο χρόνος μας, αλλά μας τελειώνουν τα μέλη. Mm-hmm. Έρχομαι στο σημείο 13, τα διάφορα. Υπάρχει κάτι υπό τα διάφορα. Όχι. Άρα, επόμενη συνεδρίαση στις 29 Ιανουαρίου από τις 9 το πρωί μέχρι το μεσημέρι τις 12.30. Ευχαριστώ. Ω, συγγνώμη. Ακυρώσαμε τη συνεδρίαση της 29 Ιανουαρίου από ό,τι φαίνεται. Καλό αυτό ίσως να ξεκουραστούμε και να έχουμε περισσότερη ενέργεια και άρα πιο ισχυρή παρουσία και περισσότερα μέλη παρόντα στις συνεδριάσεις. Αν πρέπει τελικά να μη συνεδριάζουμε για να μας λείψουν και να τους λείψουμε. Σας ευχαριστώ για σήμερα. Θα τα πούμε σύντομα.